So, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω σήμερα λίγο πιο αργά, γιατί μόλις έδωσα την άδεια σε κάποιον να πάει στην τουαλέτα. Πρώτου ξεκινήσουμε, θα επαναλάβω αυτό που είπα και το πρωί, όπου η προσέλευση ήταν μικρότερη. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές που μου αποστήλατε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς μου. Το έχω πει και στην πολιτική μου ομάδα ότι επέστρεψα μεν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για ολική επαναφορά. Παρ' όλα αυτά είμαι βέβαιος ότι θα με υποστηρίξετε και θα με επαναφέρετε προκειμένου να μπορέσω και εγώ να επανέλθω πλήρως στα καθήκοντά μου. Γι' αυτό και εύχομαι να έχουμε και στο μέλλον μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ πάντως θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Πάμε. Σημείο 7. Έγκριση γνωμοδότησης υπομορφή επιστολή σχετικά με αιτήσει κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση. Μιλούμε για την υπόθεση που σχετίζεται με την ε, Microsoft. Ψηφίστε παρακαλώ. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει. David Κάζα. Τρεις υπεράριθμοι του ΕΛΚ. Φλάισιχ, Είστε όλοι πολύ εργατικοί, πρέπει να παρατηρήσω. Ένας πλεονάζων Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Εγκρίνεται. Βλέπετε και το αποτέλεσμα στην οθόνη. Σημείο 8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά, Δεν είμαι πολύ σίγουρο. Πέρασαν και 8 μήνε. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για να είμαστε βέβαιοι. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, οπότε πέρασε ψηφοφορίε. 28 υπέρ, 21 κατά. 40 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ένας περισσεύει από το ΕΛΚ άλλη μια φορά. Πρέπει να ξανακάνουμε την ε, ψηφοφορία γιατί ένας ε, βουλευτής παραπάνω από το ΕΛΚ ψήφισε. Ψηφίστε ένας λιγότερο. Παρακαλώ. Ψηφίσατε. Ωραία, πέρασε τη ψηφοφορία. Υπέρ 29, κατά 18, 44 ε, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 47. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε φορές. Εγκρίνεται με 24 περί 20 κατά. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 50 καταπίπτει, οπότε περνάμε στην 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. <clears throat> Συμβαστική H, ήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική I, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην ε, τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13. Αποκινούμε την 100 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνονται. Μπατζ 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ρο, πι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 αποσύρθη, 105 και 106 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική Q, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. Όχι. 113. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 113 τώρα. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Οπότε ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 31 ε, υπέρ, 14 κατά. Συγγνώμη, φαίνεται ότι η όρασή μου δεν είναι ακόμα πολύ καλή. Δεν έχει επανέλθει πλήρω. 16 έχει καταπέσει, οπότε περνάμε στην τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας ψηφίσουμε καλύτερα. Ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπάτζ 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπάτζ 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 130 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, Καλύτερα να, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. 132 ψηφίστε παρακαλώ. άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. ...27 υπέρ, 23 κατά, οπότε εγκρίνεται και περνάμε... Ναι, παρακαλώ. Ψηφίσαμε την 21, τροπολογία 21, ίσως ε, το χάσαμε, την προσπεράσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Με βοηθάτε. Οπότε, πάμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και με αυτό περνάμε στην τροπολογία 133. Όχι, όχι, καταπίπτει αφού εγκρίθηκε η 132. Καταπίπτει η 133. Λοιπόν, 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136. Ε, καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβαστική 6 χ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τρεπεραλογία 22 υπέρ κατά με την 144 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι 145 ψηφίστε παρακαλώ τώρα για την τροπολογία 145 αριστη ψηφοφορία ψήφισαν όλοι ωραία οπότε ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία 30 υπέρ 19 κάτι πρέπει να κάνουμε την ώρα σήμερα 146 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται θέλει κάποιο έλεγχο ωραία τότε να το ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 146 ε, παρακαλώ ψηφίστε ψήφισαν όλοι 27 υπέρ 23 κατά κάπως βελτιώνεται η όραση μπατ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Μαζί με την 148 ταυτίζονται αυτές οι δύο τροπολογίες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Κατέπεσε συμβαστική C. Παρακαλώ πείτε μου. Να ελέγξουμε την τροπολογία 29. Ωραία. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 29 τότε. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της Εγκρίνετε. Εγκρίνεται. Οι δύο καταπίπτει. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά δεν έχω πολύ καλή εικόνα. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ζητώ συγγνώμη. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 33. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρας φοβορίες. 30 υπέρ 19 κατά. Θα προτιμούσα αν μπορούσατε λίγο περισσότερο να σηκώνετε το χέρι σας για να σας βλέπω καλύτερα. Badge 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Απεσύρθη. Μπάτς 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ για την Badge ε, 3. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Οπότε Οπότε της ψηφοφορια 25 25-25, άρα απορρίπτεται. Δίκιο είχα. Συμβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 καταπίπτει. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία σχετικά με, την, με το σχέδιο έκθεσης. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. υπέρ της ψηφοφορίας. 46 υπέρ, 3 κατά. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ίδιο ακριβώ το αποτέλεσμα. Ξανά συγχαρητήρια. Στον εισηγητή. Λοιπόν. Σημείο 9. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Συμβαστική D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 41 γιατί ίσως το πήγα πολύ γρήγορα, δεν ήταν πολύ σαφής η εικόνα. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τεροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καλύτερα να ψηφίσουμε όμως ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 44 ηλεκτρονικά τώρα. Alle τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 45-46 κατά καταπίπτει, απασύρθηκαν μάλλον, συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην badge 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σίγουρα καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρασε ψηφοφορία λοιπόν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52 με προφορική τροπολογία του Εμίλιαν Πάβελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν κατάλαβα, αν, αν το είδα σωστά. Θέλει κάποιος να ελέγξουμε? Ωραία, καλύτερα να το ελέγξουμε. Συμφωνώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε. Ωραία. Πέρας προφορία, εγκρίνεται. Τροπολογία 55 και μπάτζ 7 πρώτο τμήμα που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 απεσύρθη, συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 και μπάτζ 7 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 συμβαστική ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα συμβαστική Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 53, καλά τα λέω. sorry, sorry, K. Βαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική εμ μη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική νη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική x υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα λοιπόν. 91. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσαν όλοι. Ωραία. Τέλος της Πράγματι απορρίπτεται. Τροπολογία 93 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T. ΤΑΦ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. U, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. V, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. W, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Υ. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπάτζε 9 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά επειδή δεν είμαστε... Όχι, είμαι βέβαιος, εγκρίνεται. Συμβαστική Ζ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 με προφορική τροπολογία του Πάβελ, υπέρ, κατά, αποχές, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Μπατζ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, 129 και μπάτζ 11 ταυτίζονται υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, εποχές... δεν είναι καθόλου σαφές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 130. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, 24 κατά. 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλει κάποιος να το ελέγξουμε. Ωραία, ας το ελέγξουμε λοιπόν. Να ψηφίσουμε για την τροπολογία 138. Τώρα, ένας ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πράγματι απορρίπτεται. Ε, συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. ποχέ, Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά εποχές καλύτερα να το ελέγξουμε. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 απεσύρθη. Budget 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 37 τώρα. abgestimmt? Εγκρίνεται 28 υπέρ 23 κατά. Δύο ψηφοφορίες απομένουν ακόμη. εντολή και σύνθεση. Ας κάνουμε πρώτα την τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα να ψηφίσουμε για την εντολή. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τις Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην συγκεκριά. 10. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωση και Εργασία. Eurofound. Συμβαστική C υπέρ. Κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D2. Καλά τα λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. D2, συμβαστική D2. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσαν όλοι. Ωραία. Τέλος. Πέρασε ψηφοφορίας. What? She gave us the wrong So, we will all remember. One point, one point, point for you. Okay. Was abstimmen? Kompromiss C stimmen wir D2. D2. D2. Ας ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 20. 28 κατά. 22 υπέρ. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπατς 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ύψιλον υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε. Για τη συμβαστική ύψιλον. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας, Εγκρίνεται. Ωραία, και πρέπει να στην τροπολογία 121 υπέρ, κατά, αποχές, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 121. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της Απορρίπτεται. Συμβαστική γιώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ι2 ε, ε, μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. So, amendment 15. 15. Δεκαπέντε και μπάτζ 6 τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική κάπα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. N2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όμικρον υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Π υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Q υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. R υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. W υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 134 υπέρ Παρακαλώ. Α, όχι, ναι, καταπίπτει, έχετε δίκιο. Συμβαστική S υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 ήρθε, 129, 29 ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 κατά πίπτη. Τη 145 υπέρ κατά εποχές 145 Ψηφίσαμε για την 145 και εγκρίνεται. 146 καταπίπτει. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. U2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μπράβο, προσέχετε. Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 135 καταπίπτη και περνάμε στην 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονικά καλύτερα για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ για την 161 ηλεκτρονικά. της προφορίας και απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά όμως. 33 και 162 που ταυτίζονται υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική V2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλύτερα όμως να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να το ελέγξουμε, να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Με μικρή διαφορά απορρίπτεται. 164-165 που ταυτίζονται και 166. Και οι τρεις τροπολογίες αυτές υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνονται. Μπάτζ 8 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική χ υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Μπάτζ 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ο, καλύτερα να, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, εντάξει. Μπατζ 9. Ψηφίσατε όλοι. Συγγνώμη. Συμβαστική ζήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 κατέπεσε 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Sind wir bei 39? 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε γιατί όχι ψηφίστε παρακαλώ Alle Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 180. Όχι, κατέπεσε. Συμβαστική ΑΑ. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. 41. Απεσύρθη. Όχι, να ψηφίσουμε. 41 και 185 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. ΒΒ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θέλετε να ψηφίσουμε. Όχι, να μην ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τι θέλετε, να, να, να ελέγξουμε ή να μην ελέγξουμε. Ένα από τα δύο. Ωραία. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 41-185. Ψηφίστε τώρα παρακαλώ. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. <laughs> As long as. Uh... okay. Compromise BB. Συμβαστική ΒΒ υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 καταπίπτει, 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, δεν καταφέρα να το δω. Νομίζω ότι οι σοσιαλιστές δεν σηκώνουν αρκετά καλά τα χέρια τους. Παρακαλώ, λίγο πιο ψηλά για να βλέπουμε. Ωραία, τότε πάμε κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί όχι. Θα σας πετύχω όμως, πού θα μου πάτε. Ψηφίσατε όλοι. 198. Ψηφίσαμε όλοι. Ωραία, απορρίπτεται. 199. Περ. Κατά. Πω, πολύ δύσκολα. Πάμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Μη παραδεκτή. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις 48. Ψηφίστε. Ένας ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Κλείνουμε τη ψηφοφορία. 49 υπέρ κατά εποχές τι να πω τώρα Ωραία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για τη 49 ψηφίστε παρακαλώ. Alle abgestimmt. ist abgelehnt. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 ε, όχι καταπίπτει. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 57 ηλεκτρονικά τώρα. 2. Εγκρίνεται. Budget 2. Υπέρ κατά να το ξανακάνουμε λίγο διανατάσεως. Υπέρ, μπάτς 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 58. Απεσύρθη συμβαστική Β2. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β3 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 59 καταπίπτει. Ωραία, οπότε περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της ε, έκθεσης. ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Ψηφίσατε όλοι. Συγχαρητήρια. Στον εισηγητή. Και να ψηφίσουμε και για την εντολή. Δεύτερη ψηφοφορία λοιπόν. Ονομαστικά, ηλεκτρονικά. Τι. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τελειώσαμε και αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή και σε όλη την ομάδα του. Τελειώσαμε και με αυτή την έκθεση. Αύριο θα συζητήσουμε για σύσταση των συντονιστών. Περιμένετε, περιμένετε. Αργά, αργά. Αύριο. Ήταν μια παρατήρηση δική μου. Θα συζητήσουμε αύριο στους συντονιστές αν οι εισηγητές των τελευταίων τριών ε, εκθέσεων θα διαπραγματευτούν από κοινού. Απόφαση των συντονιστών θα είναι αυτό. Εγώ απλά είπα ότι θα το θέσουμε. Το 11 αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου και περνάμε φυσικά στον David Κάζα και το σημείο 12 της Μερισσίας Διάταξης Θεμητά μέτρα για τους ε, καταγγέλτες. Παράγραφος 1, τροπολογία 41 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το δούμε όμως και ηλεκτρονικά να είμαστε 100% σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ ένα χρησιμοφορέας. Ωραία, αν ψήφισαν όλοι τη Εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ Την M την κάναμε μόλις. Έχουμε περάσει στην επόμενη. P. Λατινικό υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Εν. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Απο, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Οκ. Okay. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 84. Ψηφίστε παρακαλώ, έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Απορρίπτεται. Συμβαστική R. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική S. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστ... Όχι. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H, με συγχωρείτε. I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σίγουρα θέλετε αλήθεια να το, να το επαληθεύσουμε. Φυσικά, φυσικά εννοείται. Αφού εκφράζεται αμφιβολίε, α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε για την τροπολογία 37. Ψηφίσατε όλοι. Amendment 38. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, όχι εντάξει, πλάκα έκανε. 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε για την ε, έκθεση στο σύνολό τη. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε και το αποτέλεσμα. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα της προφορίας. Θα πιούμε ένα προσέκο μαζί για τη μεγάλη σου επιτυχία. Σε ένα βάθαμα, σύνδευα Wer ist das? Wer ist da da? So. Wir unterbrechen mal ganz... Ωραία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Παρακαλώ. Με ακούτε. Συγγνώμη. Λοιπόν, όχι, δεν θα κάνουμε μικρό διαλυματάκι. Γιατί είναι εδώ ο προσκεκλημένος μας. Οπότε περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Και για το σκοπό αυτό καλωσορίζω ορίζω τους εκπροσώπους. Hm?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 soweit? Ready? Please take your seats. Καθίστε παρακαλώ, γιατί είμαστε έτοιμοι. Σας παρακαλώ ησυχία. Anne Sander. Felin. Feline. Ist das zu fassen? δεν το πιστεύω. Παρακαλώ δεν με ακούτε. Λοιπόν, σημείο 13. Εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Και χαιρετίζω τον Γιάννη Τιμόφσκι από το EPRS που θα μας παρουσιάσει τις, ε, τα βασικά πορίσματα της ε, αξιολόγησης, της μελέτης. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank Um, thank you very much, Chair. And... ευχαριστώ πολύ. Με χαρά το EPRS παρουσιάζει τα προϊόντα του, τα οποία αποβλέπουν στο να σας βοηθήσουν με τη δουλειά σας. Στα πέντε λεπτά και με κάποιες διαφάνειες που έχω, θα προσπαθήσω να συνοψίσω σύντομα μια δημοσίευση που έχουμε και που έχετε λάβει, ελπίζω όλοι, μέχρι τώρα. Εκεί ΓΑΜΑ και η Ερευνητική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου και μονάδα αξιολογήσεων έχουν μεταξύ άλλων στόχων την παροχή πραγματογνωμοσύνης όταν προετοιμάζεται προετοιμάζονται στάσεις όπως τώρα από την Επιτροπή μας. Με αυτή την δημοσίευση για επικαστές δύο μήνες από τη Γραμματεία επειδή όταν ξεκίνησε δουλειά το Μάρτη δεν ήμασταν σε θέση τότε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Χρησιμοποίησα τις πληροφορίες που έδωσε η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου στη συνέχεια και οι απαντές της Κομισιόν χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουμε όχι μόνο την κατάσταση σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, αλλά για να κάνουμε και κάποια αξιολόγηση του κατά πόσο επιτέχθησαν οι στόχοι και κατά πόσο αυτή η αξιολόγηση έχει περιορισμούς λόγω ακριβώς θερυψής δεδομένων. Βεβαίω, δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω και πολύ τι γίνεται εδώ με τις βασικές πληροφορίες, δηλαδή και το κατά πόσο διαβάζει το κοινό της εκθέσεις μας. Πάντως είναι σημαντικό να υπογραμμίσω το υπόβαθρο σε σχέση με τη δημοσίευση αυτή, επειδή είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των εγγυήσεων και της πρωτοβουλία για τους νέους, ιδιαίτερα στις χώρες με την υψηλότερη ενεργεία. Η πρωτοβουλία για τους νέους είναι ένα επιπλέον χρηματοοικονομικό εργαλείο και νομίζω είναι η αντίδραση της Ένωσης σε μια κατάσταση κρίσης που αποδείχθηκε μέσω αυτής ακριβώς της πρωτοβουλίας και της προχρηματοδότησης των αντίστοιχων πρωτοβουλειών. Υπάρχει και μια σχετικά περίπλοκη διαδικασία και μηχανισμός εποπτείας, σύμφωνα βέβαια και με τον κανονισμό του ECF, και προσπαθήσαμε να δούμε για ποιο λόγο η Κομισιόν δεν μπόρεσε να λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται από τις χώρες μέλη λόγω ακριβώς καθυστέρησης στην εφαρμογή των λειτουργικών των πυριακών συγγνώμη προγραμμάτων που χρειάζονται και πράγματι τα δεδομένα που μας έδωσε η Κομισιόν δεν τηρούν, δεν πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις σχέση με την υποπτία, το monitoring, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων πρέπει να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό εργαλείο της Ένωσης που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Λόγω ακριβώς του ευρύτερου πλαισίου του οικονομικού πολιτικού. Για τα δεδομένα και αυτά που αναφέρονται στη δημοσίευση καταδεικνύουν κυρίως τη δομή της εγγύησης Υπάρχει χωριστό τμήμα γι' αυτό, αλλά είναι σημαντικό αυτό το πλαίσιο να το αναφέρω. Έχουμε επίση τα επιχειρησιακά προγράμματα που ανέφερα προηγουμένω, όπου οι περισσότερε χώρε τα διαθέτουν μέχρι τώρα και η διαδικασία αποδοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αποτέλεσε έναν παράγοντα για την περαιτέρω ή τη μετέπειτα υιοθέτηση. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου τα δεδομένα για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δείχτες δεν υπάρχουν ακόμα και στην έκθεση της Κομισιόν είδαμε μια προσπάθεια για βελτίωση. Είδαμε από τους αριθμούς από τη μια μεριά την αυξημένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος και αφετέρου δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν πως σε κάποιες χώρες μέλη ο το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί. Κάτι το οποίο βέβαια είναι θετικό. Αλλά βέβαια εμείς στην έρευνά μας δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Είναι πιθανόν αυτό να έχει κάποιο αντίκτυπο όσον αφορά δηλαδή το πρόγραμμα και την πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων και την υποχώρηση τη μείωση της ανεργίας. Αλλά ομολογώ ότι δεν ξέρουμε ακριβώς αν υπάρχει άμεσος συσχετισμός ή όχι. Και στο τέλος της δημοσίευσή μας θα δείτε τις μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα στοιχεία στοιχεία του 15 και εν μέρη του 16. Οπότε σε δύο μήνες από τώρα θα έχετε μια πιο επικαιροποιημένη κατάσταση που θα μας επιτρέψει να πούμε κατά πόσο έχουν αλλάξει πολύ αυτά τα ποσοστά ή όχι. η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις προσδοκίες τώρα, εκτός από το πρόβλημα του θεσμικού πλαισίου, γιατί ήδη κάποιες χώρες διαθέτουν προηγμένο σύστημα μηχανισμών για την απασχόληση των νέων, άλλες όχι, και βέβαια αυτές οι χώρες που έχουν ευρέως χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία για τους νέους, αυτοί οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για μεμονωμένα προγράμματα, όχι για αυτά τα δομημένα προγράμματα του ESF που, όπως ξέρετε, παρεμβαίνει. Τώρα το ελεκτικό συνέδριο έθεσε ένα ζήτημα και ξέρω ότι θέλετε να το εξετάσετε, είναι το κατά πόσο η εθνική πορεία αντικαταστάθηκαν από την κοινωτική χρηματοδότηση, όχι από ό,τι φαίνεται, και κατά πόσο ο πραγματικός αντίκτυπος εδώ μπορεί να υπολογιστεί. Αυτά σχετικά με τη δημοσίευσή μας που σας καλώ να τη διαβάσετε. Είναι αρκετά δύσκολο πάντως στο σημείο αυτό να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας για τους νέους. Θα έπρεπε να ήταν πάντως ευκολότερο να γίνει κάτι τέτοιο με τα νέα δεδομένα, πάντως από ό,τι, από ό,τι γνωρίζετε υπήρξε αντίκτυπος, όχι τόσο φιλόδοξος όσο θα θέλαμε, αλλά υπάρχει. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ θα μπορούσε αυτό να ήταν χρήσιμο. Αλλά η διαφορά μεταξύ της φιλόδοξης και της δραστικής ε, προσέγγισης οδηγεί καμιά φορά σε παρανοήσεις. Και το αναφέρουμε στη σελίδα την τελευταία ότι φέτος οι δημοσιεύσεις σχολιάζοντας τις εκθέσεις της Κομισιόν λέμε ότι παρά την πρωτοβουλία παραμένει σημαντικός αριθμός ανέργων μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Αυτό σε σχέση με τους πολύ φιλόδοξους και υψηλούς στόχους για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των εργασιακών των νέων. Και ξέρετε, το συνέδριο ζήτησε από τα, θεσμα... από τα συγγνώμη, θεσμικά όργανα της Ένωσης να επιδείξουν ρεαλισμό για αυτά τα θέματα ώστε να είμαστε επιτυχείς. Αυτά από μένα σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή. Την εισηγητρία, αν Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης με την εμπειρογνωμοσύνη τους συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτού του σχέδιου έκθεσης γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτό το έργο κατανοήσαμε γρήγορα ότι δεν θα ήταν εύκολο για όλους τους λόγους που αναφέραμε. Έχουμε πολύ λίγα δηλαδή ε, στοιχεία ποιοτικά σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, καταφέραμε να προετοιμάσουμε και να διατυπώσουμε κάποια μηνύματα κλειδιά, τα οποία ε, περιλαμβάνονται επίση σε αυτή την έκθεση και αντικατοπτρίζουν και την ε, άποψή μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας τα εκθέσω με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θέσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή ποιο είναι το μέλλον αυτής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ε, Το κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και πώς είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ε, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την αποστολή μας. Ε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ποσοστό ανεργίας εξαιρετικά ψηλό για τους νέους και αυτοί οι νέοι ελπίζω ότι θα μπορέσουν να βασιστούν στη δική μας βοήθεια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό ε, σε αυτή την υπόθεση είναι τι θα πρέπει να γίνει με αυτά τα χρήματα που έχουν χορηγηθεί για αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να αυξηθεί το κονδύλι. Εγώ πιστεύω πως ναι και το στηρίζω αυτό, αλλά θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε ο προπολογισμό αυτός να εκτελεστεί με υπεύθυνο τρόπο, πιο υπεύθυνο από ό,τι μέχρι τώρα. Στην έκθεση αυτή υπογράμμισα επίσης την σημασία της πολιτικής θέλησης και της πολιτικής στήριξης. Όταν δηλαδή μιλάμε για την ανεργία των νέων, που είναι επίσης πολύ σημαντική, και επίσης να τονίσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Πιστεύω πως οι νέοι ξεκινούν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δεν οδηγούν οπωσδήποτε στην ε, εργασία. Άρα χρειάζεται αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα γιατί μπορεί πάντοτε να ρίχνουμε χρήματα αλλά παραμένουν ε, βραχυπρόθεσμα αυτά τα μέτρα και οδηγούν σε μια τεχνητή δημιουργία θέσεων. Εμείς θα θέλαμε οι θέσεις αυτές να είναι πιο βιώσιμες, πιο διαρκείας. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τον ίδιο τον ορισμό της ποιοτική προσφοράς θέσεων απασχόλησης, γιατί πρόκειται για έναν τομέα όπου δεν έχουμε βρει συμφωνία. Όταν όμως ε, μελετούμε διαφορετικές πηγές, ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι θέσεις απασχόλησης οι οποίες δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων συνήθως έχουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα αλλά και τη διάρκεια τους. Γιατί μια θέση που για παράδειγμα διαρκεί μόλις κάποιους μήνες ή θέσεις οι οποίες δεν είναι καλής ποιότητας δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ικανοποιητικέ ως αποτέλεσμα το να αυξηθεί η ηλικία στα 29 έτη νομίζω είναι πολύ καλή απόφαση διότι οι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας όσο, ε, όσο πάει και αργότερα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση γι' αυτό και ε, το συγκεκριμένο είναι μέτρο το οποίο θεωρώ πολύ θετικό. Και για να κλείσω θα ήθελα επίσης να τονίσω, να υπογραμμίσω ένα θέμα που σχετίζεται με το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, ποια περιοχή, ποια περιφέρεια θα πάρει αυτά τα κονδύλια, ίσως θα ήταν ε, σκόπεμο να χορηγηθούν αυτοί οι πόροι σε μικρότερες περιφέρειες από τις σημερινές, γιατί εγώ είμαι πεπισμένη ότι μια αναδιοργάνωση σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή θα μας επέτρεπε να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα και να συμβάλλουμε έτσι στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα αυτού του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας μια αποστολή επιτόπου 19 με 21 Σεπτεμβρίου και θα επισκεφθούμε δύο χώρες, τη Σλοβενία και την Κροατία, ε, αποστολή που θα μας επιτρέψει να συναντήσουμε φορείς ε, επιτόπου Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε πολλά σημαντικά πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Είστε όλοι λοιπόν ευπρόσδεκτοι και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας εύχομαι δε καλές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπενιφέη για τους σοσιαλιστές. Grazie ευχαριστώ ευχαριστώ την Συγχύτρια για την παρουσίαση του σχεδίου. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε μεταξύ μας εμείς οι σκιώδεις. Δεν είναι η πρώτη ανταλλαγή. Και πρέπει να πω ότι είχε ανοιχτή η διάθεση η από την αρχή. Να πω ότι σε σχέση με τους λομπίστες που συναντήσαμε το περασμένο μήνα, ήταν απαραίτητο να έχουμε κάποιες παρατηρήσεις και σε σχέση με εκείνη τη συνάντηση νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος εργασίας, δηλαδή τακτικά να τα λέμε μαζί τους και στις μετέπειτα φάσεις της εργασίας της, της Επιτροπής μετά από την αποστολή βέβαια στην Κροατία και την Σλοβενία. Δεν είναι μόνο θέμα μεθόδου, αλλά σημαντική πολιτική επιλογή. Μα ε, προσφέρει την ευκαιρία η έκθεση αυτή να κάνουμε όχι μόνο τεχνική αλλά και πολιτική δουλειά και να ανυψώσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου σε θέματα που αφορούν πρωτοβουλίε για την απασχόληση των νέων και τι εγγύησει. Οπότε συμμερίζουμε αυτά που είπε η συγγήτρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έγγραφο για να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών σε σχέση με τους στόχους των εγγύσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις συστάσεις για τη μελλοντική βελτίωση. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι και από τα κρισιμότερα που είδαμε επαλημένως σε διάφορες χώρες φέτος η ποιότητα εργασίας που προσφέρεται στους νέους και αυτό αφορά και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που αποδεικνύει, αποδεικνύεται χρήσιμη στο να επικριθούν προγράμματα τα οποία αποδεικνύονται αναποτελεσματικά σε σχέση με τους πόρους που χρησιμοποιούνται ή την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τους νέους ανενεργούς εργασιακά. Μας δείχνει όμως και άλλα στοιχεία, όπως ας πούμε για τη δουλειά της Κομισιόν και τη μελέτη που έγινε για την απασχόληση των νέων στη ΣΥΠΑ όπως ακριβώς ε, λέγει η έκθεση της Κομισιόν πέρσι. Τώρα για το θέμα της ποιότητας λοιπόν της προσφοράς εργασίας. Αυτό είναι ένα ακριβές παράδειγμα του πώς εμείς θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να προωθούμε παγκόσμιες αξίες όσον αφορά την ποιότητα της προσφοράς εργασίας. Και η Κομισιόν και ο παγκόσμιο Οργανισμός Εργασίας και το Συμβούλιο ακριβώς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το θέμα της προσφοράς εργασίας. Ως ένα θέμα που αφορά ακριβώς το, τα προσόντα των νέων και την προσφορά, αλλά αυτό από μόνο του είναι περιοριστικό. Και νομίζω πάντως για τα πολιτικά θα βρούμε κάποια συμφωνία οι πολιτικές ομάδες. Χαίρομαι επίση που η συγκίτρια αναφέρεται επίση στου πόρου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την απασχόληση των νέων, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί την πρώτη βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Και τέλος, συμμερίζομαι την ανάλυση ότι οι πρωτοβουλίε και οι εγγύησεις θα πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία για τη διευκόλυνση τη λεπτή φάση μετάβαση προ πλήρη απασχόληση. Αλλά από μόνα του δεν μπορούν να προκαλέσουν ε, εργασία, θέσεις εργασίας. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε φιλόδοξε ευρωπαϊκέ πολιτικέ που θα αποβλέπουν στην προώθηση και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίστηκε με λαθασμένες συνταγές μακροοικονομικής πολιτικής και είχαν αντίκτυπο δραματικό στους πιο ευάλωτους, θα πρέπει να αλλάξουμε βιβατισμό και θα πρέπει να πάμε σε επενδύσεις στα κοινωνικά θέματα. Και θεωρώ ακριβώς λοιπόν ότι οι εγγύσεις των νέων και οι πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων θα μπορούσαν να αποδειχτούν χρήσιμα εργαλεία για την διευκόλυνση αυτής της σημαντικής δουλειάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη Γκέρικε, εκ μέρους της ηγήτριας για το ECR. Έχει το λόγο. Would κοιόδης μας εισηγητρία θέλει να ευχαριστήσει την εισηγητρία και τους κοιόδης εισηγητές. Πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση όπου εργαζόμαστε περισσότερο με συνένεση και η ομάδα μας είναι ευτυχής που το κείμενο αντικατοπτρίζει αυτά που θεωρούμε σημαντικά. Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι, σημαντική είναι η σταθερή και ισχυρή προσπάθεια και δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών, έτσι ώστε να λειτουργήσει η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και να έχει αυτά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα για μα εξαρτώνται από τη βιώσιμη απασχόληση. Μαζί με τους κοιόδη εισηγητέ, νομίζω πω έχουμε επίση στήριξη για καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη βελτίωσή του στο μέλλον, καθώ και στην προσαρμογή του στι ανάγκε των νέων νέων. Επίσης, ε, με χαροποίησε που είδα στο κείμενο μία έκκληση για μεγαλύτερη επαφή με τους νέους που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασία, για παράδειγμα νέου με ε, ειδικέ ανάγκε. Προσβλέπω στην ε, εργασία, εργασία αυτή και στηρίζω την αρχική εκτίμηση τη εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω εκ μέρου τη δική μα εισηγήτρια. Ματίνα Κύριε για το Άλτε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την για την ε, συνάντηση των σκιωδών των ε, εμπλεκομένων φορέων. Είδαμε την έκθεση, είδαμε τα δεδομένα. Δεν κατάφερα όμω να τα διαβάσω στην ε, την παρουσίαση αυτή. Δεν, την έβλεπα καλά από την οθόνη. Ίσως θα μπορούσατε να μας την εκτυπώσετε, να μας την αποστείλετε μάλλον, για να έχουμε μια βάση συζήτησης. Στις μελλοντικές ε, συναντήσεις των συντονιστών νομίζω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά, γιατί στην έκθεση, και ο Ρωμάνα το έκανε ήδη αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τόσο τα θετικά που βγήκαν από την πρωτοβουλία, αλλά και τα μειονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον. Ε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτές τις αδυναμίες. Για παράδειγμα είναι το μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής της πρωτοβουλίας, δυσκολίες προσδιορισμού των πραγματικών αναγκών, διοικητικό γραφειοκρατικό άχθος που εμπόδισαν την πρόοδο του συστήματος, του, της πρωτοβουλίας, απουσία αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, ποιότητα των προσφορών, κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, προσπάθειες των κρατών μελών για την καλύτερη διασύνδεση των εκπαιδευτικών συστημάτων με την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα ε, αποτελούν ένα τρίγωνο. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να συμμετέχουν η αγορά εργασία, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι φορεί χάραξη πολιτική. Όλε αυτέ οι τρει ε, περιπλέψει θα πρέπει να συνεργαστούν. Όχι μόνο σε μια οριζόντια συνεργασία, αλλά και σε μια κάθετη συνεργασία. Γιατί χρειαζόμαστε συμπράξει μεταξύ διαφόρων επιπέδων της διοίκησης, ε, ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού, τοπικού επίπεδου. Αυτά είναι νομίζω τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Και ε, νομίζω ότι δηλωτικό του γεγονότος ότι η συζήτηση αυτή είναι όρημη είναι και το γεγονός ότι συμμετέχουν και όλες οι άλλες επιτροπές με γνωμοδοτήσεις είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουμε ε, γνωμοδότηση των Επιτροπών Προϋπολογισμού, ε, το, της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που ελέγχει βεβαίω και την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος. Εν πάση περιπτώσει προσβλέπω σε αυτήν την συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξαιρετικά ισορροπημένη προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κονσάλε για την ε, ΓΚΟΕ. Ε- Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Τάνκ για τη δουλειά της. Έχω κάποιες κατευθυντικές γραμμές που θα τα κάνω να δουλέψουμε πάνω σε αυτές και νομίζω είναι σημαντικό να εξολογήσουμε τα αποτρέσματα αυτής της πρωτοβουλίας για τους νέους μετά από πέντε χρόνια έχουμε επίπεδα ανησυχητικά για το 20% της ε, ανεργίας των νέων και για την χώρα μου είμαστε πάνω από το 40% χώρα μου την Ισπανία. Και βλέποντας την έκθεση του Ολεκτικού Συνεδρίου καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρξε συνεννόηση πανευρωπαϊκή, ο καθένας υιοθέτησε τα δικά του μέτρα. Υπάρχουν χώρες που χρησιμοποίησαν τα κονδύλια για να κάνουν προγράμματα μέσω φορέων περιφερειακών ή επαγγελματικών σε άλλες χώρες. Είχαμε μια αντικατάσταση των ε, πολιτικών απασχόλησης σε εθνική κλίμακα. Και με τον ίδιο τρόπο ο μηχανισμός χρηματοδότησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου δεν βοήθησε τη ταχεία υλοποίηση προγραμμάτων για τις χώρες που τα χρειαζόταν περισσότερο παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ως επιτυχία το γεγονός ότι 14 εκατομμύρια εργαζόμενοι ε, εντάχθηκαν στις εγγυήσει και 3 εκατομμύρια στην πρωτοβουλία για την απασχόληση, ε, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ζήτησης, αλλά προσφοράς και ποιότητας της εργασίας. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι αυτό. Και νομίζω ότι όταν σχεδιάστηκε η εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας αυτής για τους νέους, δεν έλαβα υπόψη τους και τόσο το θέμα της έλλειψης των ευκαιριών, αντί για την απασχολησιμότητα. Οι ευκαιρίες λοιπόν. Και αυτό που βλέπουμε σε πολλές χώρες είναι ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, βραχύβιες, προσωρινές, απασχόλησης, με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Οπότε πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση η οποία ακριβώς θα πρέπει να μεταμορφώνει και να προωθεί την απασχόληση που δεν υπάρχει μέσω κοινοτόμων προγραμμάτων που θα αξιοποιούν ακριβώς τα νέα ταλέντα και θα προωθούν μορφές κοινωνικής οικονομίας. Δηλαδή σε τελική ανάλυση μας λείπουν πρωτοβουλίες ακριβώς που θα δημιουργήσουν την απασχόληση που λείπει, όχι που θα διαμορφώσουν την υπάρξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον για το έγγραφο αυτό που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησής μας. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο μηνύματα που νομίζω ότι υπάρχει συνένεση γύρω από αυτά και αυτή είναι και η βάση της έκθεσης. Πρώτον, θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτή την πρωτοβουλία, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα και δεύτερον ότι θέλουμε να λύσουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν γιατί φυσικά όλοι έχουμε σε μια κριτική στα οποία μπορούμε να ασκήσουμε Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν ορισμένα ε, σημεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν για να γίνει πιο ολοκληρωμένο, να, να καταργηθούν ορισμένε διακρίσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που τα ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Πρώτον, πράγματι, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια πολύ καλή αξιολόγηση τη κατάσταση, γιατί δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα επαρκή δεδομένα. Και νομίζω ότι αυτό θα, θα, θα δυσκολέψει το έργο για την σύνταξη αυτής της έκθεσης. Παρ' όλα αυτά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεύτερον, ε, αυτό που ανέφερε και ο εισηγητής, πώς ακριβώς ε, ε, ορίζει κανείς το θέμα της ποιότητας. Είναι και πολιτικό το θέμα αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία επισφαλών ε, θέσεων μέσω αυτής της πρωτοβουλίας ε, και νομίζω και κάτι ακόμη που μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο είναι ότι από την εμπειρία μας ε, γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά στέφθηκαν πάντοτε με επιτυχία όταν υπήρχε συμμετοχή και των νέων οργανώσεων των, των νέων των ιδίων δηλαδή ανθρώπων στα οποία απευθύνονται αυτά τα προγράμματα και νομίζω ότι αυτό καλό θα είναι να ε, αναφέρεται ρητά στα, στην έκθεση και νομίζω ότι εδώ ως Κοινοβούλιο έχουμε πραγματικά αποδείξει το γεγονός ότι μας νοιάζει η συμμετοχή των ε, νέων ανθρώπων. Έχουμε κάνει μεγάλες συζητήσεις, έχουμε κάνει διερευνητικές αποστολές, έχουμε έρθει σε επαφή με οργανώσεις των νέων και νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν για να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Μέλα από το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Η προηγούμενη έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των νέων λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαπιστώνει ότι σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εκτιμήσει τον αριθμό των νέων που έχουν ε, ε, εποφεληθεί από αυτά τα προγράμματα για την απασχόληση των νέων. Γι' αυτό και ζητά την εφαρμογή των εισεγγύησης για τους νέους και την πρωτοβουλία αυτή για τους νέους ε, ώστε να έχει συγκρίσιμα στοιχεία επιτέλους Επιπλέον εκτιμά ότι υπάρχει ένας ε, σημαντικός κίνδυνος στα κονδύλια αυτά να υποκαθιστούν τα εθνικά σχετικά κονδύλια. Η συγχρηματοδότηση ζητά να είναι υποχρεωτική και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε βεβαίως. Δεν έχουμε τίποτα άλλο νέο. Ε, αρκούμαστε στο να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να διορθωθούν αυτά τα ελαττώματα, αλλά κυρίως δείχνει την ανεπάρκεια αυτής της διάταξης που λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Ε, θα, επίσης τίθεται το ερώτημα πού πήγαν αυτά τα χρήματα που έχουν επενδυθεί σε αυτό το πρόγραμμα μέχρι στιγμής να μην περιμένουμε πολλά για να μπορέσουμε να κρίνουμε τα επιτόπου αποτελέσματα και πρέπει να το πούμε η ενεργεία των νέων είναι μία από τις μεγάλες αποτυχίες της ευρωπαϊκής πολιτικής και όλος ιδιαιτέρως σε θέματα απασχόλησης να θυμίσουμε ότι 20 με 25% των νέων κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι και για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και θα συμμετέχουμε επιμελώς σε αυτήν την συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει χρόνος και για άλλες παρεμβάσεις αν θέλετε, αλλά πέραν του εισηγητή και των ε, σχεδόν δεν βλέπω κάποιον. Α, είναι η Ντανούτα. Ντανούτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. με που δεν με είδατε νωρίτερα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρωμάνα για την γνωμοδότησή της, την, την έκθεσή της. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να, συναντήσουμε τους ανθρώπους στους, ε, ε, στον τόπο τους για να δούμε τι πράγματι έχει επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι είναι ε, πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να διοργανώνει τέτοιου είδου συναντήσει. Έγινε και μάλιστα μια τέτοια συνάντηση με χορηγό τον κύριο Μπάλας για την κοινωνική ασφάλιση με τη συμμετοχή διαφόρων οργανώσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Πρέπει πραγματικά να, να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους ε, στους οποίους απευθύνονται αυτά τα προγράμματα και για τους οποίους έχουν ε, αναπτυχθεί. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αναφορές από το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με την πρωτοβουλία για τους νέους και την απασχόληση των νέων. Και εξακολουθούμε να ακούμε διαρκώς για αδυναμίες και προβλήματα ή λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε ε, αν τα χρήματα αυτών των προγραμμάτων δαπανώνται σωστά και αν έχουν τελικά και κανένα σοβαρό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε όμως να συλλέξουμε ε, κάποια στοιχεία. Χι εκατομμύρια νέοι εκπαιδεύτηκαν και ψι εκατομμύρια άνθρωποι, νέοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Όχι για τρεις μήνες, κανονική δουλειά, μακροπρόθεσμη να δούμε αν η εκπαίδευση αντιστοιχεί στις ανάγκες των εργοδοτών. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Οι δάσκαλοι στις χώρες μας, οι καθηγητές, δεν ε, ε, συμβαδίζουν με τις αλλαγές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας ή με, τα, με τις αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα. Να εκπαιδεύουμε ανθρώπους να στέλνουν βιογραφικά ή να φτιάχνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα διοικούνται στη βάση της συναπόφασης. Όποιος συμμετέχει δηλαδή, συμμετέχει και στη λήψη των αποφάσεων. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζονται και επενδύσει στο εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να λειτουργήσουν ω μέντορε. Δεν αρκεί απλώ να λειτουργούν ως ημάντες μεταφορά γνώσεων. Πρέπει να εξηγούν οι εκπαιδευτικοί στου νέου ανθρώπου για το πώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τι πληροφορίε και όχι απλά να τι απορροφήσουν στατικά. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω να πετύχουμε στη διαδικασία αυτή διότι σε τελική ανάλυση νομίζω ότι ε, αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να δρέψουμε και τους καρπούς αυτών των προγραμμάτων. Η εγγύηση για τους νέους και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μάλιστα θα μπορούσαν και να συγχωνευτούν διότι έχουν και, οι δύο πολύ θετικές, και τα δύο πολύ θετικές πλευρές. Θυμάμαι ότι η κυρία Σαρτιά και ο κύριος Ρόιντεν ε, μας πήγαν στις ε, περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου, των κατοχωρών, της Γαλλία, όπου και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με νέους ανθρώπους για τις εγγύησει για τους νέους, για παράδειγμα. Οπότε και μας είπαν ότι δεν θέλουμε, ε, δεν θέλουμε εγγύησεις για του νέους, δουλειέ θέλουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ντανούτα, συγγνώμη που δεν σε είχα δει. Άλλε παρεμβάσει. Ωραία, τότε να κάνω και εγώ τρεις παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως ε, ε, κίνητρα για την συνέχιση της συζήτησης. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Εγώ ως ε, συμμετέχων στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία έχω ζήσει η διοίκηση ε, στη Γερμανία να προσπαθεί με διάφορα στατιστικά μέτρα να, να αντιμετωπίσει την ανεργία χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Διότι αποκλειστικός σκοπός ήταν να μειωθεί ο αριθμός, το ποσοστό της ανεργίας. Αν μέσω αυτών των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών υπηρετείται κάποιος τέτοιος στόχος, τότε νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, διότι η πραγματική ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στα δικά μας μέσα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε βοήθεια για αυτοβοήθεια. Με άλλα λόγια, να βοηθήσουμε ε, τα εθνικά κράτη-μέλη να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα. Τρίτον, αν θέλουμε να συζητήσουμε για ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα ισχυρότερο από το πακέτο Juncker, το οποίο θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, τότε αυτό, για, για κάτι τέτοιο, δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε μόνο στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τέλος, κάτι που το απευθύνω κυρίως προς την Κομισιόν, αλλά μπορούν να το σκεφτούν και οι σκιώδεις. Νομίζω ότι η επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη έχει ένα, ε, ε, παρουσιάζει πανευρωπαϊκά πολύ μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την ποιότητά της. Γι' αυτό... Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Ντανούτα για, την, ε, για τις δυνατότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών. Δηλαδή, να μην δίνουμε απλά νέες πληροφορίες και γνώσεις στους νέους, αλλά να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Διότι πολύ συχνά ακούμε και από συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και από τους εργοδότες ότι η εκπαίδευση έχει μείνει 10 χρόνια πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά, ε, με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και χρειάζεται να δουλέψουμε και πάνω στον τομέα των ε, εκπαιδευτών. Και νομίζω ότι αν χαράξουμε μια τέτοια κατεύθυνση εδώ στο Επιτροπή Απασχόλησης, θα καταστήσουμε και αυτά τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες πιο αποτελεσματικές. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή όλων σε αυτή τη συζήτηση και αυτή τη διαδικασία. 26 ε, Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου για τις τροπολογίες αυτές και ε, από εκεί και πέρα θα γίνει και η ψηφοφορία στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Πότε θα πάει στην Ολομία δεν ξέρουμε ακόμα. Παρ' όλα αυτά είναι βέβαιο ότι έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς μπροστά μας. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει ο καιρός. Σας ευχαριστώ πάντως για την συνεργασία σας. Και με αυτό περνάμε στο τελευταίο σημείο της σα διάταξης. Πολύ πολύ πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε αρχικώς. Είναι εδώ η συντάκτρια γνωμοδότησης μεν, όμως δεν είναι εδώ η σκιώδης. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα ή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν και πολλά με ένα μικρό διαλυματάκι. Η Σοφία Ριμπέρο δεν είναι εδώ. Μαρία Ρέινα επίσης δεν είναι εδώ. Α, εδώ είναι, όχι, λάθος έκανα. Μαρία, πώ ήταν δυνατόν να μη εδώ. δω. και Τριμπέζιου, Μπόιλεν, Λίπουν, Τάμας Μέζαριτ, επίση δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι. Ωραία, πάμε να περάσουμε στο θέμα. Σημείο Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ, Γιάννα Τόμ, σχέδιο της Έχετε το λόγο, Γιάννα. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω γιατί έχουν φύγει οι Είναι σχεδόν η τελευταία μέρα εργασιών. Μπορώ να τους σας στείλω και γραπτός από εκεί και πέρα και νομίζω ότι έτσι κι η συνεργασία μας θα είναι πάρα πολύ καλή. Συνάδελφοι, να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για τις οικονομικές πολιτικές ζώνες του ευρώ. Πρώτα θα σας δώσω κάποια ε, ε, στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια θετικά νέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Τον Μάρτιο του 2017 πήγε στο 9,7 ε, η ανεργία. Είναι θετική δυναμική, ωστόσο στις αρχές του 2016 ήταν 10,2. Παρά τις θετικές εξελίξεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν επανέλθει στα επίπεδα προκρίση. Οι ανησυχίε μου επίση σχετίζονται με την ε, νεανική ανεργία. Συμφωνώ με αυτό που έχετε πει στις ε, καταληκτικές σας παρατηρήσεις στην, ε, στην προηγούμενη εισηγήτρια, αλλά για μας είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ζήτημα η ανεργία των νέων. Τον Μάρτιο ε, η ανεργία των ε, νέων ανερχόταν σε 19,4, χαμηλότερη από ότι πέρσι 22 περίπου τις 100, παρόλα αυτά είναι απαράδεκτα υψηλή ακόμη. Βρίζεται ότι τα κράτη-μέλη ε, έχουν πολύ μεγάλη διαφορέ όσον αφορά τις αποδόσεις των αγορών εργασίας τους. Σε κάποιο βαθμό η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έχουν καθυστερήσει και ε, παρά, το γεγονός ότι ε, εκδόθηκαν ε, συστάσεις αναχώρα. Ε, πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες να αυξηθούν. Επίσης πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να εξασφαλίσει απαραίτητα κονδύλια για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία αυτής της πρωτοβουλίας έπειτα από τα πρόσφατα ευρήματα του Ελληνικού Συνεδρίου την ειδική έκθεση για την ελληνική ανεργία. Η έκθεση αυτή λέει ότι κανένα από τα κράτη-μέλη δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει όλοι οι νέοι άνθρωποι που δεν βρίσκονται στην εργασία, την απασχόληση ή την κατάρτιση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία πρόσφορα με μορφή που θα τους βοηθήσει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με βιώσιμο και ε, διαρκή τρόπο. Καθώς ε, η νομοθεσία για τις εγγύσεις για τους νέους ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη, πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη αυτά. Η γαλλική ανεργία πολλές φορές είναι αποτέλεσμα αποτυχία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η ανεπαρκώς χρηματοδοτηθήσα εκπαίδευση πολλές φορές υποσκάπτει τις αγοράς εργασίας, τις αγοράς εργασίας μέσω της ανυπαρξίας ε, επαρκών ε, ατόμων με τα απαραίτητα προσόντα. Ε, η νεανική ανεργία ε, σε πολλά κράτη-μέλη έχει μειωθεί. Φυσικά αυτό το ζήτημα, ιδίως στην οικονομική του διάσταση, είναι ε, θέμα και αρμοδιότητα άλλης επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν θα πρέπει να υπάρχει μια στενή ερμηνεία της, ε, το, το, της ψηφιακής ε, εκπαίδευσης με το να χρησιμοποιούνται δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες πλατφόρμες. Η απουσία αυτών των ε, προσόντων και δεξιοτήτων υποσκάπτει ακόμη και τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Νομίζω ότι τα επόμενα δέκα χρόνια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στην αγορά εργασίας αν δεν έχεις ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης είναι σημαντική η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Επίσης χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να ε, εξασφαλιστεί η ισορροπία τη οικονομικής και της κοινωνικής διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί αυτό θα βελτιώσει συνολικά την οικονομική κατάσταση. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ε, φτώχειας των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική κατά τη φτώχεια για να επιτευχθούν στόχοι για το 2020. Επίση, πρέπει να δίνονται ισχυρότερε ε, συστάσει στα κράτη-μέλη για την κοινωνική συνοχή και ένταξη. Και νομίζω ότι μπορούν τα συστήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση τη φτώχεια. Αυτέ είναι κάποιε από τι παρατηρήσει και σκέψει μου και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα για να ακούσω και τι δικέ σας απόψει. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε μαζί μα μόνο μία σκιώδη, την Μαρία Ρένα από τους Σοσιαλιστέ, η οποία και εκπροσωπεί όλους τους υπόλοιπους σκιώδεις εκ των πραγμάτων. Αρένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την συγγύτρια για την παρουσίαση. Συμφωνώ με το ότι αν έχει υποχωρήσει ενεργεία χαιρόμαστε, αλλά όχι πολύ όμως, γιατί δείχνουν στατιστικές και τα στοιχεία ότι οι θέσεις αυτές δεν είναι ποιότητας. Ούτε έχει βελτιωθεί λοιπόν η ποιότητα εργασίας, ούτε η ποιότητα ζωής των πολιτών. Βλέπουν σε κάποιες περιοχές υπάρχουν μεγάλες διαφορές για την ανεργία μεταξύ χωρών και μεταξύ εσωτερικών χωρών. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές, σημαντικοί θύλακες ανεργίας και επίσης οι πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι και οι γυναίκες επειδή ακριβώς είναι υπερβολικά υψηλό το ποσοστό ανεργία των γυναικών σήμερα στην Ευρώπη και σε διάφορες περιοχές βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες για τους σοσιαλιστές ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα της κοινωνική Ευρώπης. Είπατε ότι το κυριότερο θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση που πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε ιδιαίτερα για τους νέους μας. Νέους που είναι σήμερα πτυχιούχοι αλλά άνεργοι αλλά και για αυτούς που δεν είναι πτυχιούχοι και αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πάνω στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους νέους. Την εκπαίδευση βέβαια μέσω εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και την άτυπη μέσω απασχόλησης. Όπως είπαμε, στόχος μας είναι να αυξηθούν αυτοί, αυτά τα εργαλεία για τους νέους. Επειδή δεν, δεν είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους σήμερα που είχε θεσπιστεί από την ε, Κομισιόν, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα παρατήσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά και θα πρέπει να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τους νέους και τις εγγύησεις. Μάλιστα και θα έλεγα ότι αν μπορέσουμε να υποχρεώσουμε τις χώρες μέλη να τηρήσουν ένα σύμφωνο δημοσιονομικό, τότε εξίσου θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποχρεώσουμε τις χώρες να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την ανεργία των νέων. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης και των νέων μας, οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί σε σχέση με αυτές τις εγγύσεις για τους νέους και την αποτελεσματικότητά τους. Θέλω λοιπόν περισσότερα και θέλω καλύτερα για τους νέους να κάνουμε τρίτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι πολιτική που θα προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή. Μίλησα προηγουμένω για τι αποκλήσει όσον αφορά την αργία μεταξύ των γυναικών σήμερα. Αυτό συνδέεται συχνά με την ε, αδυναμία να συνδυάσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ώστε να συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Έχουμε θέματα όπως οι αδείς πατρότητες και αλλά και πάλι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά ας πούμε, την υποδοχή των παιδιών και άλλες υπηρεσίες που θα επιτρέψουν να συγκεράσουμε τις δύο ζωές. Η επόμενη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για κάποιους τα συνδικάτα θεωρούνται ως εμπόδια επειδή ακριβώς προστατεύουν τους εργαζόμενους βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι ένα μοντέλο ισορροπίας πρόσβασης στις δυνάμεις αυτές, τις συνδικαλιστικές ε, και τις εργοδοτικές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας λείπουν εργαλεία ισορροπίας σε σχέση με αυτές τις δύο δυνάμεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν η Ένωση μέσω διαλόγου να ενισχύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ώστε να έχουμε συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους οι οποίες θα τους αρμόζουν καλύτερα. Και ιδιαίτερα βέβαια οι συλλογικές συμβάσεις έχουν τεράστια σημασία. Αλλά μια πρωτοβουλία που συμβαδίζει με τον κοινωνικό διάλογο είναι η ενίσχυση των συνεταιριστικών δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της πόλωσης των αμοιβών, κάτι το οποίο σήμερα είναι έντονο φαινόμενο στην Ευρώπη. Η ενίσχυση επίσης των συστηματοκοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου πυλώνα, πυλώνα των συντάξεων, αλλά και του πυλώνα υγείας. Είδαμε κατά τη διάρκεια του τριμήνου του Ευρωπαϊκού ότι οι συστάσεις αναχώρα της Κομισιόν είναι συστάσεις οι οποίες ευνοούν την ιδιωτικοποίηση αυτών των πυλώνων, δηλαδή η ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα των συντάξεων και εξασθενεί, εξα, εξ, αποδυναμώνει τον πρώτο πυλώνα που είναι ο πιο ισότιμος και που αφορά τις συντάξεις για τους ε, εργαζόμενους και για τους εργαζόμενους η απόκληση στις συντάξεις μεταξύ αδών και γυναικών ξυπνά το 40% στην Ευρώπη. Αν λοιπόν παραβλέψουμε τον πρώτο πυλώνα και ενισχύσουμε τον δεύτερο και τον τρίτο, τότε αυτοί αποκλείσαν ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί οι γυναίκε σήμερα εργάζονται στην Ευρώπη στου φτωχούς κλάδους της οικονομίας, που δεν συμβάλλουν πολύ σε αυτού τους πυλώνες τη σύνταξη. Σε σχέση δηλαδή με το δεύτερο και το τρίτο που είναι ιδιωτικέ συντάξει. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τον την πρόνοια. Και πρόεδρε, μια και με μόνη μου θα τα πω όλα εγώ. Πρέπει να βελτιώσουμε βεβαίω τι ε, συνθήκε εργασία, το είπαμε αυτό, την ποιότητά του, Θα αυτό σε σχέση με την προσωρινή εργασία, αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και το κοινωνικό dumping. Δηλαδή, αυτό το φαινόμενο που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και αυτές οι πρακτικές που το συνοδεύουν καταστρέφουν την εξέλιξη της ευημερία των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις, τις αφαιρεσίες στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι απαραίτητο αυτό για να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα οι πολίτες. Επίσης χρειαζόμαστε κοινωνικού δείκτες. Κοινωνικούς δείκτες, γιατί αν θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά τα μέτρα που λαμβάνουμε θα πρέπει να έχουμε σωστούς δείκτες επίσης. Και βαρέθηκα πια να μιλάμε για το ΑΕΠ συνέχεια, ΑΕΠ και ΑΕΠ και ΑΕΠ και ανάπτυξη Ήρθε η ώρα να έχουμε σωστούς δείκτες κοινωνικούς, προσμετρήσιμους, υπολογίσιμους, που θα έχουν την ίδια αξία με τους καθαρά οικονομικούς δείκτες. Ευχαριστώ. So, dann danke ich den mindestens, dann danke... Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν τους πέντε σκιώδεις που μόλις πήραν το λόγο. Για το EFDD δεν υπάρχει σκιώδης, ούτε για το ENF. Δεν βλέπω κάποιος άλλο να ζητά το λόγο λοιπόν. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορούμε να τελειώσουμε για σήμερα. Προθεσμία για τροπολογίες είναι 19 εβδόμου. 16 λένε τα έγγραφά μου, αλλά δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό. Οπότε στις 12 το μεσημέρι, στις 19... 28 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε το θέμα. Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την ΕΚΟΝ και στις 16 Οκτωβρίου θα, θα ψηφίσει η ΕΚΟΝ για την γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και τελειώνοντας πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε ε, προβλέψει. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Hmm?